να σας ενημερώσω ότι ο κύριος Ροζάριο Κροτσέτα, πρώην βουλευτής του Κοινοβουλίου, απίφθινε στον Πρόεδρο αίτηση για την πράσπιση της βουλευτικής του ασυλίας στα πλαίσια μιας προδικαστικής διαδικασίας στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο του Παλέρμο. Βάσει του κανονισμού αποστέλλεται στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου το θέμα, η οποία είναι και καθήλυνα αρμόδια. Περνάμε τώρα στις ψηφοφορίες.